περνάμε στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας. Ευχαριστώ πολύ. Συνεδρίαση ΙΜΚΟ, ε, στην οποία βεβαίως μπορούν να παραμείνουν και τα μέλη της Επιτροπής Γιούρι, αν θέλουν να μας πούν ε, την, ε, τις δικές τους γνώμες. μιλούμε για τις συμβάσεις, για την για τις ηλεκτρονικές και άλλες εξαποστάσεις πωλήσει αγαθών. Και θα δώσω το λόγο κατευθείαν στον κύριο Σαμπμάιερ για να παρουσιάσει την πρόταση και τη μελέτη αντικτύπου για, για τις ηλεκτρονικές και άλλες εξαποστάσεις πωλήσης αγαθών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Um, as we... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή έχουμε ε, ξεπεράσει το χρόνο μας πολύ σύντομα. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι σε συνδυασμό με την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο πρόκειται για ένα από τα πρώτα παραδοτέα στην, ε, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Έχουν εντοπιστεί ορισμένα προβλήματα και γι' αυτό η Κομισιόν του επόμενους μήνες θα προτείνει διάφορες δράσεις. Εδώ όμως ε, διαπιστώσαμε ότι ένα από τα βασικότερα εμπόδια για την ψηφιακή ενιαία αγορά ε, σχετίζεται με το δίκαιο περισυμβάσεων. Και αυτό για τους καταναλωτές συμβαίνει την ε, συμβατότητα, την ε, μη παροχή ή την παροχή εσφαλμένου ε, αγαθού και γι' αυτό σχετίζεται το ζήτημα αυτό με τα ένδικα μέσα. Για τις επιχειρήσεις ε, πρόβλημα είναι ε, γενικά οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών κτλ. Δεν θα σας δώσω πολλά στοιχεία. Βασικά αυτό που βρήκαμε ήταν ότι μόνο ένα μικρό μέρος των καταναλωτών 38% συγκεκριμένα, νιώθουν εμπιστοσύνη για να αγοράσουν ηλεκτρονικά από άλλη χώρα. Τρεις, ε, από τις βασικότερες ανησυχίες είναι τι θα συμβεί αν ε, υπάρχει κάποιο σφάλμα, θα υπάρχει επισκευή, αντικατάσταση, τι γίνεται με την ε, επιστροφή των χρημάτων και τι γίνεται με τα ελαττωματικά προϊόντα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς με την πρόταση είναι να παράσχουμε ορισμένα ωφέλη για τους καταναλωτές με την μορφή της μεγαλύτερης ποικιλία επιλογής και την, των χαμηλότερων τιμών και ε, όλα αυτά με, βεβαίως με δεδομένο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών. Για τις επιχειρήσεις οι διαφορές ε, στα, μεταξύ των εθνικών δικαίων είναι πολύ σημαντικές ακόμα και για το 40% των επιχειρήσεων που ήδη ε, συναλλάσσονται διασυνοριακά. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να παράσχουμε στις επιχειρήσεις είναι το εξής. Ένα κοινό σύνολο κανόνων στη βάση του οποίου θα μπορούσαν να πουλήσουν τα αγαθά τους, τα προϊόντα τους σε όλες τις χώρες της ενιαίας αγοράς. Και αυτό θα οδηγούσε, αν υπήρχαν δηλαδή οι ίδιοι κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 57% των ε, επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινούσαν ή τουλάχιστον θα εξέταζαν την πιθανότητα να πουλήσουν ε, τα προϊόντα τους διασυνοριακά. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι η διάκριση μεταξύ ε, των κανόνων για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το παραδοσιακό εμπόριο. Είπα και εισαγωγικά για την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο ε, ότι ένα από τα βασικά αποτελέσματα της διαβούλευσης ήταν ότι οι άνθρωποι μας είπαν ότι αν εναρμονίσετε το ψηφιακό περιεχόμενο και προσπαθήσετε να ε, ευθυγραμμιστείτε όσο το δυνατόν περισσότερο με, τις, ε, με το καθεστώς για τις ηλεκτρονικές πωλήσει, αυτό εμεί αυτό εμείς θα το θέλαμε. Το κάναμε. Αν όμως εναρμονίσουμε τους κανόνες για τις ε, ηλεκτρονικές πωλήσει, τότε θα πρέπει να εναρμονιστούν και οι κανόνες ε, των ε, παραδοσιακών πωλήσεων. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε τα απαραίτητα δεδομένα για να κάνουμε μια τέτοια πρόταση. Και μιας και διακηρύσουμε την καλύτερη νομοθεσία, θα πρέπει και να καταλήγουμε σε αντίστοιχα αποτελέσματα. Και επειδή έχει ήδη προγραμματιστεί η διαδικασία refit, έχουμε ήδη ε, ε, εξετάσει το, το ζήτημα. Ε, συλλέγουμε αυτή τη στιγμή δεδομένα, θα, θα τα έχουμε έτοιμα τον Ιούλιο ε, για αυτό το θέμα και το σκεπτικό μας ήταν ότι μόλις συλλέξουμε τα απαραίτητα δεδομένα θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε στο τέλος να έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο κανόνων για όλες τις πωλήσει. Γιατί ακολουθήσαμε αυτήν την οδό. Διότι θεωρήσαμε ότι ε, είναι σωστό να ξεκινήσουμε με την ψηφιακή διάσταση των πολίσεων. Υπήρχε ε, συνένεση ότι το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να ρυθμιστεί γρήγορα. Αν δεν το κάνουμε θα χάσουμε το τρένο αλλά το ψηφιακό περιεχόμενο από μόνο του ε, αφορά συγκεκριμένες μερίδες των εμπορικών συναλλαγών, ε, ένα μικρό μέρος των εμπορικών συναλλαγών. Αυξανόμενο σίγουρα, αλλά πάντως μικρό ακόμη. Αν θέλουμε εμείς να επιτύχουμε την ανάπτυξη, ε, δεν θα την επιτύχουμε μόνο μέσω του ψηφιακού περιεχομένου και γι' αυτό ήταν σημαντικό να έχουμε και την ψηφιακή διάσταση και γι' αυτό κάναμε τα πράγματα όπως τα κάναμε. Και επιπλέον, από τη διαβούλευσή μας το προηγούμενο καλοκαίρι και με όλε τις συζητήσει με κράτη-μέλη και ενδιαφερόμενου, θεωρούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα καλύψαμε όλα τα ζητήματα που είναι κοινά και για τις ε, online και για τις offline πωλήσει. Ε, ενδεχομένως υπάρχουν κάποια ζητήματα που σχετίζονται μόνο με τις παραδοσιακέ πωλήσει, τις μη επιγραμμικέ δηλαδή, αλλά νομίζουμε ότι αναδείξαμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Κομισιόν στην ανακοίνωσή τη. Ε, δεσμεύτηκε ότι θέλουμε ως στρατηγικό στόχο να επιτύχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο κανόνων. Και για αυτό το σκοπό θα αξιοποιήσουμε και τα δεδομένα που θα συλλέξουμε. Για την πρόταση, πάρα πολύ σύντομα θα σας τα πω. Υπάρχουν τρεις βασικές ουσιώδεις τάσεις στην πρόταση αυτή. Πρώτον, η πρώτη ουσιώδη στάση είναι ότι επιμένουμε στα ζητήματα που ρυθμίζονται στην ε, οδηγία για τις πωλήσει. Να ε, εντοπίζουμε συγκεκριμένα διασυνορικά προβλήματα και να υπάρχει και συνέπεια με την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και γι' αυτό το λόγο η πρότασή μας ρυθμίζει ε, κατά κύριο λόγο τα ένδικα μέσα, τη δοκιμή συμβατότητας και, τα, και τις αποζημιώσεις. Επίσης, αυξάνουμε το επίπεδο προστασίας καταναλωτών σε σύγκριση με την οδηγία για τις ε, πωλήσει προς καταναλωτές. Και το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το βάρος απόδειξης αυξάνεται από 6 μήνες σε 2 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την προστασία των καταναλωτών και πρόκειται για αύξηση της περίοδου, της προβλεπόμενης περίοδου για τις 26 από τις 28 χώρες. Επίσης, ε, η πρόταση ε, αφαιρεί την υποχρέωση από τον καταναλωτή να κοινοποιεί το πρόβλημα στον πάροχο. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα λύσης της σύμβασης λόγω μη συμβατότητας, ακόμη και αν το ελάττωμα είναι ε, έλασον και επίσης υπάρχουν ε, λιγότερες ε, περίοδοι εγγύησης για μεταχειρισμένα προϊόντα και τέλος υπάρχουν απλούστεροι ε, κανόνες για να περάσει ένας καταναλωτής από, το πρώτο επίπεδο ένδικων μέσων στο δεύτερο επίπεδο ένδικων μέσων. Άρα αυξάνουμε σημαντικά την προστασία των καταναλωτών και τέλος η τελευταία τάση είναι ότι εμείς ε, χρησιμοποίησαμε και διατύπωση η οποία προσωμιάζει προς εκείνη της οδηγίας για τις πωλήσει και πρόκειται για διατύπωση που έχει υιοθετήσει και το Κοινοβούλιο σε διάφορες τροπολογίες και στους, στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Χρησιμοποιούμε δηλαδή ε, μια πιο σύγχρονη ορολογία από ότι αυτή της οδηγίας του 99. Σε τελική ανάλυση όμως επιμένουμε και επικεντρώνουμε στα βασικά προβλήματα και μια μετάβαση από την προηγούμενη προσέγγιση. Πρόκειται για μια πρόταση με στόχο την πλήρη εναρμόνιση που αντιμετωπίζει τα κοινά προβλήματα που θέλει να αυξήσει το επίπεδο εμπιστοσύνη από την, των, των καταναλωτών αφενό και αφετέρου να διευκολύνει τι επιχειρήσει να πολλούν τα αγαθά του διασυνοριακά. Ευχαριστώ. οι συζητητέ ε, τη ΣΥΜΚΟ πρώτα και δεν ξέρω αν θέλει κανένα άλλο ε, να πάρει το λόγο. Πασκάλ Αριμών πρώτο που είναι εισηγητή και μετά η Λούση Άντερσον. Evelyn Gephardt, Angel Cecilia Wikström, Yuri Mestalka, Joel Bergeron. Um, μερικοί είναι εκτός, μερικοί είναι απόντες, ε, θα ξανάρθουν, εν πάση περιπτώσει. Αυτή ήταν η σκέψη. Καλώς. Ο Πασκάλα Ευχαριστώ, Βίκη. Καταρχάς, εισαγωγικά. Σε σχέση με την πρώτη της οδηγίας, εγώ είμαι ε, ένθερμος υποστηριξής πλήρους εναρμόνισης. Αυτό είναι καλό και για την προστασία των καταναλωτών, αλλά και για εκείνους που κάνουν επιγραμμικό εμπόριο. Αλλά δεν είμαι ο μόνος εδώ υπέρ ε, της πλήρους εναρμόνισης, ούτε ε, και πεπισμένος ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να πείσουμε τους πάντες ότι αυτό είναι κάτι καλό. Ορισμένοι διαφωνούν και κυρίως στο Συμβούλιο. Κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν πιστεί. Και αυτή η μελέτη αντικτύπου, μεταξύ άλλων, έχει και αυτό το σκοπό να βρούμε επιχειρήματα για να πείσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Εξού και η σημερινή ακρόαση που είναι τμήμα αυτής της δουλειάς που πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ τώρα ψάχνω επιχειρήματα έτσι ώστε το κείμενο αυτό με αυτή τη μορφή ή με κάποια αλλαγή μικρή στη διατύπωση να ευδοκιμήσει και να επιτύχει. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό είναι καλό και για το εμπόριο και για τους καταναλωτές. Ε, οπότε, έχω έξι ερωτήσεις για να μου δοθούν απαντήσεις και θετικά επιχειρήματα να πείσω και εκείνους που δυσπιστούν. Πρώτον, υπάρχουν ήδη δύο οδηγίες οι οποίε τώρα γίνονται τέσσερι. Οδηγία σημαίνει ότι το κράτο μέρο θα πρέπει να την εφαρμόσει, να τη μεταφέρει στην νομοθεσία και δεν είναι απόλυτη εναρμόνιση αυτό. Υπάρχει οδηγία το 1999 για ε, ε, τις αγορές ε, των προϊόντων ή του 2011 για την προστασία των καταναλωτών και έρχονται να προσθεθούν άλλες δύο προτάσεις. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μήπως έχετε σκεφτεί αντί να τις κάνετε τέσσερις να τις κάνετε μία, τις δύο αυτές οδηγίες ή τις δύο παλαιότερες απλώς να τις συμπληρώσετε για λόγους έτσι ε, απλότητας. Το δεύτερο που με βασανίζει και που θα μπορούσε να είναι και ένα σημείο τριβή, είναι η σημερινή διάκριση που γίνεται σε αγορέ επιγραμμικές και μη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαφορά αν παραμείνει έτσι. σχέση με το τι δικαιούμαι ως ε, παροχές για προϊόντα, αν πάω να αγοράσω κάτι σε ένα μαγαζί ή το αγοράσω από τον υπολογιστή μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγηλε ότι την οδηγία του 99 στη ε, διαδικασία REFIT την αναθεωρεί και την εξετάζει. Και ρωτώ συγκεκριμένα, έχετε κάποια ενδιάμεσα αποτελέσματα και πότε μπορούμε να περιμένουμε τα τελικά. Επίσης, Τι προτιμάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από εκεί και πέρα να κάνει. Προσανατολίζεστε σε αλλαγή της υφιστάμενης πρότασης της οδηγίας ή θα κάνετε μια τελείως νέα πρόταση. Γιατί δεν θα πάμε από τις 2 στις 4 αλλά από τις 2 στις 5. Έτσι πώς το βλέπετε πιο πρακτικά να γίνεται και πιο απλά. Τρίτη ερώτηση. Η εκτίμηση των επιπτώσεων του αντικτύπου impact assessment της οδηγίας. Εδώ λέει ότι αν έχουμε πλήρη εναρμόνιση, αυτό σημαίνει 0,03% αύξηση του ετησίου ε, κύκλου εργασιών, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια. Αυτά τα έχετε μελετήσει και για την εναρμόνιση, αν γινόταν εξίσου για τις επιγραμμικές και μη επιγραμμικές πωλήσει. Αν εναρμονίσουμε τα πάντα, δεν θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Τέταρτο, έρχομαι ακριβώς στα επίμαχα σημεία στην πρόταση αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, τώρα είναι μια εξαιτία και προτείνεται διετία. Για τον καταναλωτή αυτό είναι φανταστικό, αλλά για τον λιανέμπορο μάλλον όχι. Πρώτον, ρωτήσατε τους εμπόρους και τι λένε. Είναι ευτυχείς, χαίρονται γι' αυτό τους ικανοποιεί και από την απάντησή σας πραγματικά θέλω να λύσω επιχειρήματα για να μπορώ να πείσω τους εμπόρους ότι είναι καλό ή και τα κρατημέλη που εκπροσωπούν. Και έρχομαι στη διετή ε, προθεσμία για την εγγύηση των δικαιωμάτων. Αυτή η πρόταση που εναρμονίζει τα πάντα δίνει τη δυνατότητα προθεσμιών στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν να μειώσουν την προστασία των καταναλωτών. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο, α πούμε, αυτή τη στιγμή κιόλα είναι πολύ ε, ευαίσθητο το θέμα, αλλά εκτό του Ηνωμένου Βασιλείου είναι και η Φιλανδία και η Ιρλανδία και κάτω χώρε που μειώνουν την προθεσμία αυτή. Ε, στο Βέλγιο και στην Γαλλία ε, ε, υπάρχει η έννοια του vis κασέ που είναι η κρυφή ε, βλάβη. Είναι μια, μια, ένα ελάττωμα ας πούμε που δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Τι γίνεται με αυτό. Auf die zwei Jahre im Artikel 8.3 ist, glaube ich, so, dass As... Αν υπάρχει μια βαρύ, ας πούμε, κάποιες χώρες που έχουν μεγαλύτερες ε, διάρκειες ε, προστασίας των καταναλωτών και των δικαιωμάτων τους δεν είναι σε μειονεκτική θέση. Το έχετε συζητήσει αυτό με τους ε, ενεχομένους και τους ενδιαφερομένους στα κράτη-μέλη. Για να υπάρξει μια ισορροπία. Γιατί στην αντιστροφή του βάρους απόδειξης που περνάμε από την εξαετία στη διετία και την εναρμόνιση της εξασφάλισης της προστασίας των καταναλωτών για μια διετία, αυτό είναι θετικό ή οι χώρες τώρα που μειώνουν αυτές τις προθεσμίες συμφωνούν. Οι διαπραγματεύσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και αυτή η, η, ε, σε 13 κράτη-μέλη ε, δεν ισχύει για μεταχειρισμένα αγαθά. Ε, ε, ισχύει ένα έτος, το οποίο ένα θα γίνεται δύο. Δηλαδή, αν αγοράσω επιγραμμικά τώρα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, ε, θα έχω ε, κάλυψη για τα δικαιώματά μου ένα χρόνο ή δύο. Δεν το διάβασα στη μελέτη αντικτύπου, αλλά αυτό είναι σημαντικό κλάδο στην ευρωπαϊκή ε, οικονομία. Το έχετε συζητήσει μαζί του. Και το έχετε συζητήσει και με εκείνου που κάνουν κανονικό εμπόριο μεταχειρισμένο, α πούμε, αυτό ο ένα χρόνο να γίνει δύο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, Λουσί Άντερσον. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με κάποιε από τι ανησυχίε που ανέφερε ο συνάδελφο από το ΕΛΚΑ, αλλά πρέπει να πω εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ότι εμεί το βλέπουμε λίγο διαφορετικά Πρόφανώς ε, συμφωνούμε με το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς αγαθών ε, και συμφωνούμε με τα καλύτερα δικαιώματα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όντως βελτιώνουμε, ότι δεν βελτιώνουμε τα δικαιώματα των πολυεθνικών εταιριών ε, σε σχέση με τους απλούς καταναλωτές. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε να άρξει μια σωστή ισορροπία για όλους. Γι' αυτό νομίζω ότι η αρχή της πλήρους εναρμόνισης ε, ε, δεν, νομίζω ότι πρέπει να επιφυλαχθούμε για αυτήν την αρχή, για τους λόγους που ανέφερε και ο συνάδελφος. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε στην ε, αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και οι επιλογές που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το μέτρο ε, αυτό χρήζουν περισσότερης προσοχής. Εγώ ε, θα ήθελα να... Ε, ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλάβει, να καταλάβει τις ανησυχίες μας αυτές και γιατί κάποιες, κάποια δικαιώματα ε, βελτιώνονται και άλλα όχι. Ε, πού ακριβώς έγινε η διαφορά για τις μικρές ε, επιχειρήσεις ή για τους καταναλωτές. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εμπόδια, τα σημαντικά στο δίκαιο των συμβάσεων. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ε, νιώθουν ότι είναι διαφορετικό ε, το δίκαιο σε κάθε χώρα και ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε αυτό που κάνουν. Αν δει κανείς τα τεχνικά παραρτήματα, ε, είναι πολύ μικρό το δείγμα των επιχειρήσεων που έχει χρησιμοποιηθεί και που έχουν ερωτηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού είναι τα αποδεικτικά στοιχεία. Πάρα πολύ καλό είναι ε, να επενδυμίσουμε επίση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όταν κάποιο ε, κηρύσει καλύτερη νομοθεσία, πρέπει να προβαίνει και ο ίδιο σε καλύτερε προτάσει νομοθεσία. Για κάποια άλλα σημεία τώρα. Γιατί να διαλύξουμε το ένα και όχι το άλλο. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δικαίωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το δικαίωμα υπαναχώρηση σε μία σύμβαση, αν ε, είναι λατωματικό ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Αλλά για να το κάνουμε αυτό ε, αν δεν το κάνουμε αυτό, ε, μας, μας λέτε ότι πρέπει να υπάρχει κάποια αποζημίωση, κάποια επα, επανόρθωση. Δεν να σας πω κάτι όμως. Καθημερινή του ζωή, οι άνθρωποι δεν έχουν τον χρόνο να κάνουν αυτή τη δουλειά να πιάνουν τώρα κουβεντούλα με τον Λιανοπολιτή, αν κάτι μπορεί να φτιαχτεί ή όχι. Αν δεν δουλεύει, να το στείλουμε πίσω και τελείωσε. Και μας το λένε αυτό οι ενώσεις καταναλωτών όσον αφορά την εξαετή περίοδο περιορισμού. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και αναφέρθηκε και προηγουμένως γιατί αυτό είναι η παναχώρηση. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο συμβιβασμό ω προ αυτό. Γιατί μιλήσατε για το να πείσουμε κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Η ιδέα της μέγιστης, της μέγιστης δεν θα περάσει. Όσον αφορά την αποζημίωση, θα ήθελα περισσότερες αποσαφηνήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί από ό,τι κατάλαβα, παρά την εναρμόνιση και την προσέγγιση αυτή, θα υπάρχει μια ευελιξία σε σχέση με, τις, ε, με την αποζημίωση σε εθνικό επίπεδο. Εμείς έχουμε ότι στο Ηνωμένο, στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένο τρόπο, υπάρχουν άλλε επιλογέ ε, ε, σε κάποιε άλλε κράτη ε, χώρες μέλη, θα υπάρξουν ευελιξίες γύρω από τις αποζημιώσεις. Όσον αφορά τώρα την ε, αντιστροφή του άχθους απόδειξης, καλό είναι αυτό, αλλά αν ρωτήσετε ενός καταναλωτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πόσο σημαντικό είναι, για παράδειγμα, αυτό, αυτή η αντιστροφή του ε, άχθους απόδειξης, πόσο σημαντική είναι, αν μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στο βραχυπρόθεσμο δικαίωμα απόρριψης ενός ελαττωματικού προϊόντος ή ε, του, του δικαιώματος αυτού, ε, να σας πω την αλήθεια, ξέρω τι θα διάλεγα, θα διάλεγαν το πρώτο. Έχουμε πάρα πολλές φορές ε, συζητήσει αυτό το θέμα της καλύτερης νομοθεσίας σε αυτό το πλαίσιο. Χρειαζόμαστε περισσότερα αποδεκτικά στοιχεία γιατί κάποιες εναλλακτικές επιλογές δεν ελήφθησαν υπόψη. Για ποιο λόγο, που είναι αποδεκτικά στοιχεία, υπάρχουν τεράστιες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, οι οποίε μπορεί να μα βοηθήσουν πάρα πολύ, γιατί δεν θα μα ε, δώσουν όλα τα λεπτομερή στοιχεία που χρειαζόμαστε. Όσον αφορά την ολοκλήρωση του συμβολέου ε, λόγω ε, ελαττωμάτων, μπορεί να μην θέλουμε να επιλέξουμε αυτή την οδό, μπορεί να θέλουμε να επιλέξουμε κάτι άλλο. Όταν πηγαίνει κανείς σε ένα μαγαζί να αγοράσει κάτι, ένας απλός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο αν κάποιος αγοράσει κάτι ηλεκτρονικά, ε, Συγγνώμη, θα ολοκληρώσω, αλλά με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Αν αγοράσει κάποιος κάτι ηλεκτρονικά, έχει λιγότερα δικαιώματα από ότι αν πάει να το βγάλει από ένα ράφι σε ένα μαγαζί. Ε, επίσης το θέμα των εκ του νόμου δικαιωμάτων. Ε, εμείς δεν θέλουμε να αποκλείονται αυτά λόγω των ε, συμβατικών δικαιωμάτων. Ε, είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά είναι μόνο λίγα εξ αυτών. Ε, δεν λέω ότι δεν μπορούν να επιληθούν, ειδικότερα αν υπάρχουν συμβασμοί, αλλά η εναρμόνιση πρέπει να γίνεται προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει εναρμόνιση. Συγγνώμη, Λούση πάρα πολύ σημαντικά είναι όλα αυτά που μας είπες και πολύ καλά και πράγματι έχουν ε, θέσει πολύ σημαντικά θέματα οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά πρέπει και άλλοι συνάδελφοι να μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, συνάδελφοι, ότι εμείς ήμασταν πρωτοστάτες ε, της ε, χρήσης αξιολόγηση αξιολόγησης αντικτύπου και είπαμε μάλιστα ότι αν όλες οι αρμόδιες επιτροπές ε, θεωρούσαν ότι υπήρχαν στοιχεία τα οποία ε, δεν ε, μας κάλυπταν, θα ζητούσαμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου δική μας, όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εισηγητή έχει θέσει κάποια θέματα ω προ αυτό, οπότε ενδεχομένω και οι σκιώδει να θέλουν να το θέσουν. Πάντω, αν θέλει να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ Βίκη. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι εξηγήσει τη και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθει αυτή η πρόταση, γιατί καθημερινά αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Είναι πολύ χαμηλή η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ιδιαίτερα στο Βέλγιο, ε, όταν πρόκειται για αγορές επιγραμμικές χρειάζεται μια εξασφάλιση και επικρατεί ανασφάλεια γιατί είναι κανόνες ένα χάο πολύ διαφορετική και δεν ξέρει τελικά κατανοητή τι ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Και υπάρχουν διάφορα δίκαια ενοχικά που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ακούσαμε όμως ότι αυτό μπορεί να αυξήσει το τζίρο των εμπόρων μέχρι και 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε υπέρ της καλύτερης νομοθεσίας αλλά και της απλούστερης και της πιο εύκολης. Ε, έχω τρία σημεία να σας αναφέρω. Πρώτον, η πρόταση αυτή θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία που ήδη ισχύει. Για παράδειγμα, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και για τις, ε, την οδηγία για τις ε, πωλήσει και τις εγγύησεις για τους καταναλωτές. Θα πρέπει να προσέξουμε ε, πριν κάνουμε νέους κανόνες μήπως χρειαστεί απλώς να αναθεωρήσουμε την κείμενη νομοθεσία. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις επιγραμμικές ή τις κλασικές παραδοσιακές πωλήσει. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ένδικα μέσα, τις αποζημιώσεις λοιπά Και θέλω να ρωτήσω ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν το έχει λάβει υπόψη. Δεύτερον, η ε, ε, ε, περίοδος εγγύησης και στροφή του βάρους της απόδειξης. Χρειάζεται προσοχή να δώσουμε εδώ για να υπάρξει ισορροπία και ρεαλισμός. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να επιλέξει ο καταναλωτής επισκευή αντικατάσταση. Γιατί το επιλέξατε αυτό, γιατί το προτείνετε, γιατί ο καταναλωτής σου λέει γιατί να το φτιάξω, να μου δώσετε καινούριο. Ε, επίσης, υπάρχουν ε, κάποιες κατηγορίες ε, προϊόντων ε, ε, που μπορεί ε, κάποιο καταναλωτή να αποφασίσει μετά από μια διετία, μια τριετία ότι θέλει να το αλλάξει ε, και όχι να το φτιάξει. Και το τρίτο που θέλω να πω, να ρωτήσω δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σκέφτεστε να βάλετε κάποιες προθεσμίες με χρονικό περιορισμό. Έχαμε τώρα στο τελευταίο, έχει σημασία ε, και οι δύο προτάσεις για το ψηφιακό περιεχόμενο που συζητούσαμε προηγουμένως και ε, το τωρινό θα πρέπει να ειδωθούν ως πακέτο έτσι ώστε τα σημαντικά σημεία του ενός κειμένου να βρίσκουν αντανάκλαση ε, στο δεύτερο. Ευχαριστώ κυρία Κάλλας. Για το πεδίο εφαρμογή. Κατανοούμε όλοι ότι η Επιτροπή ήθελε να επικεντρωθεί στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Ε, αλλά ε, σκεπτόμενοι ότι δεν θέλουμε να βοηθήσουμε μόνο τις μεγάλες εταιρείες που κάνουν διασυνοριακές πωλήσει, αλλά και τις μικρές ε, επιχειρήσεις που ενδεχομένως να μην κάνουν διασυνοριακές πωλήσει, ίσως ε, θα μπορούσαν αυτές οι επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις αυτές ενδεχομένως ε, κάνουν και offline και online πωλήσεις. Και το είπε και η Λούση Άντερσον. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το ότι θα υπάρχουν δύο σύνολα κανόνων για τα υλικά αγαθά που πολλούνται στο διαδίκτυο και αυτά που πολλούνται σε παραδοσιακά καταστήματα. Ε, για την άσκηση Refit που ανέφερε η Κομισιόν, πώς η διαδικασία αυτή θα, Πώς θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία αυτή τα δεδομένα που συλλέγεται. Αν δηλαδή προχύψει από αυτή τη διαδικασία ότι ενδεχομένως χρειάζεται να γίνουν αλλαγές, θα κάνετε ε, ε, τροποποιήσεις στην πρόταση που έχετε ήδη υποβάλει, πώς θα το κάνετε. Όσον αφορά την περίοδο εγγύησης που αναφέρθηκε, και από άλλους συναδέλφους. Εγώ έχω ένα ερώτημα μόνο. Πώς λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια ζωής ενός υλικού αγαθού. Γιατί όταν σκεφτόμαστε τα σημερινά αγαθά, μπορεί αυτά πολλές φορές να μην μπορεί κανείς να τα, να μην μπορεί καν να τα χρησιμοποιήσει μετά από δύο χρόνια από τη στιγμή που τα έχει αγοράσει, γιατί έχει προχωρήσει τεχνολογία. Άρα, ε, κατά τη γνώμη μου, ε, μια τέτοια διάταξη θα έπρεπε να ισχύει για προϊόντα με μεγάλο κύκλο ζωής. Ψυγεία, για παράδειγμα. Για όλα τα υπόλοιπα, όμως, μάλλον δεν θα πρέπει να ισχύσει κάτι τέτοιο. Καταλα... Κατανοώ ότι υπάρχουν διάφοροι κανόνες σε διαφορετικά κράτη-μέλη, αλλά όσον αφορά την, την περίοδο συμβατότητας που σε κάποια κράτη-μέλη είναι δύο χρόνια και σε άλλα είναι έξι μήνες. Γιατί δίνεται αυτή την έμφαση σε αυτή την περίοδο και όχι στην περίοδο εγγύηση. Επίσης, ένα ζήτημα που ανέκυψε και στο ζήτημα του ψηφιακού περιεχομένου. Και συγγνώμη που το ξαναθέτω το ερώτημα, μάλλον δεν κατάλαβα την απάντησή σας. Έχουμε λοιπόν συνδεδεμένες συσκευές, το ίντερνετ των αντικειμένων. Η πρόταση λοιπόν λέει ότι οι κανόνες αυτοί αφορούν ψηφιακό περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο σε υλικά αγαθά. Λογισμικό ψυγείο για παράδειγμα. Από τη σκοπιά όμως του καταναλωτή, αν το ψυγείο δεν λειτουργεί, ο καταναλωτής αυτός θα πάει στο κατάστημα από το οποίο αγόρασε το, το ψυγείο και όχι σε αυτόν που ε, έφτιαξε το λογισμικό παρόλο που μπορεί το λογισμικό να είναι το πρόβλημα. Ξέρω ότι το έχετε εξηγήσει ήδη πάρα πολλές φορές και συγγνώμη που ξαναθέτω το ερώτημα, αλλά παρακαλώ ξαναεξηγήστε το μου, γιατί ε, κάποιοι ευρωβουλευτές συμπεριλαμβανομένου εμού δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς ε, την απάντησή σας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Τζούλια. Ευχαριστώ. Καταρχάς, ε, εκπλήσωμαι που από τη σκοπιά των καταναλωτών ε, ίσως ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πολύ δύσκολο να, δια, να γίνει διάκραση μεταξύ ελαττώματος ε, του hardware και ελαττώματος του software. Αλλά αυτό δεν αρκεί για να πει κανείς ότι ε, είναι σωστό να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες όταν αγοράζει κανείς ένα προϊόν online ή από παραδοσιακό κατάστημα. Ως γενική αρχή. Εμείς πιστεύουμε ότι κάθε πλήρης εναρμόνιση της νομοθεσίας για τους καταναλωτές δεν θα πρέπει να οδηγεί σε υποβάθμιση του επίπεδου προστασίας. Το είπε και η συνάδελφος από τους σοσιαλιστές. Και γι' αυτόν τον λόγο στο ψηφιακό περιεχόμενο είπαμε ότι εντάξει είναι νέος τομέας οπότε δεν θα υπάρξει υποβάθμιση της, του επίπεδου προστασίας. Αλλά εδώ είναι σαφές ότι σε κάποιες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά την περίοδο ε, εγγύησης, ναι, εδώ πραγματικά έχουμε μια ε, υποβάθμιση των ε, ισχυών των κανόνων. Και αυτό είναι θεμελιώδες πρόβλημα γιατί θα πρέπει ενδεχομένω να σκεφτούμε μήπως είναι και ένας ολισθηρός δρόμος. Αν αρχίσουμε δηλαδή να μειώνουμε τους κανόνες που ισχύουν για τις ε, ε online πωλήσει, μπορεί να καταλήξουμε τελικά και σε μείωση των κανόνων ε, για τις offline πωλήσει. Ε, και για λόγους συνεκτικότητας, γιατί υπάρχει και αυτός ο στόχος να έχουμε συνεκτικούς κανόνες. Άρα έχουμε αυτές τις ανησυχίες. Εγώ προσωπικά δηλαδή έχω αυτές τις ανησυχίες αυτές τις προτάσεις. Συμφωνούμε πραγματικά με αυτή την προσέγγιση να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές και τις παραδοσιακές πωλήσει. Νομίζω ότι μόνο αν απαντήσουμε σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα θα μπορούσαμε από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε ε, με τα επιμέρους ζητήματα της πρότασης. Αλλά πρώτα πρέπει να λυθεί αυτό. Εύελιν Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να επαναλάβω πολλά από αυτά που υπόθηκαν. Αλλά δεν θέλω να τα επαναλάβω. Να, πω όμως δύο-τρεις παρατηρήσεις που μου φαίνονται πολύ πράγματα που μου φαίνονται πολύ προβληματικά. Πρώτον αυτή η διάκραση μεταξύ online και offline πωλήσεων δεν μπορώ να την καταλάβω. Ε, αν, δείτε στο άρθρο 2 του, σύμβάση του, της σύμβασης εξ εγώ καταλαβαίνω ότι πηγαίνω σε ένα κατάστημα, βλέπω κάτι που θα ήθελα να το αγοράσω, ε, σε αυτό το κατάστημα υπάρχει ένα, ένας υπολογιστές μέσω του οποίου μπορώ να κάνω την αγορά μου. Εδώ υπάρχει φυσική παρουσία του πολιτή και του αγοραστή. Εδώ μιλάμε για offline ε, αγορά παρότι είμαι στο κατάστημα. Αν δε βγω στο πεζοδρόμιο και κάνω την αγορά από το iPhone μου, τότε ε, πρόκειται για online αγορά και θα έχω άλλα δικαιώματα από ότι αν είχα κάνει την αγορά μέσα στο κατάστημα. Είναι λίγο περίεργα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να διευθετήσουμε διάφορες λεπτομέρειες, να ξαναπεξεργαστούμε το όλο ζήτημα, γιατί είναι πολύ προβληματικό αυτό το, το σημείο. Επίσης προβληματικό θεωρώ ότι στο πλαίσιο της ελάχιστης εναρμόνισης, ε, της πλήρους εναρμόνισης, αυτά που ε, έχουμε ήδη ως κανόνες ε, ελάχιστης εναρμόνισης, αυτοί που θεσπίστηκαν πριν από δύο χρόνια δηλαδή, βλέπουμε ότι ε, στα, τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίσουν ε, περαιτέρω κανόνες ε, για τις online πωλήσει, αλλά όχι για τις offline πωλήσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και το ίδιο ισχύει και για τις προθεσμίες εγγύησης, αλλά και αυτό το δικαίωμα απόρριψης που υπάρχει στη Βρετανία αλλά όχι σε άλλες χώρες, αλλά είναι πολύ σημαντικό δικαίωμα στη χώρα αυτή. Αλλά και σε άλλους τομείς. όπως αυτή η, η ιεραρχία των αξιώσεων εγγυήσεων που επίσης ρυθμίζονται με ε, διαφορετικό τρόπο ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Στη Γερμανία υπάρχει, για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία όχι. Για ποιο λόγο όμως θα πρέπει από τους Βρετανείς να, να, να, να τους αφαιρέσουμε ένα δικαίωμα που ε, το έχουν τώρα, μέσω της πλήρους ε, ε, βλέπω εδώ διάφορα στοιχεία, διάφορε διάφορες χρόνους που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, συμφωνώ και με αυτό που είπε η κυρία Κάλλας για τη διάρκεια ζωής. Για παράδειγμα, για αυτό το μολύβι εδώ, το στυλό που σας, που δείχνω, δεν χρειάζομαι την, την ίδια περίοδο εγγύησης όπως για το πλυντήριό μου. Είναι πράγματα που πραγματικά πρέπει να τα συζητήσουμε διεξοδικά και στα οποία δεν μπορούμε απλά να πούμε ότι μπορούμε μόνο κοντιλιά να τα ρυθμίσουμε όλα. Για μένα λοιπόν ε, θα, πω το εξής. Πλήρης εναρμόνιση θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από εμένα μόνο αν υπάρχει ε, υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών όσον αφορά τα διάφορα δικαιώματα εγγυήσεις, τις αξιώσεις, ε, και διάφορα δικαιώματα που ισχύουν σε επιμέρους ε, χώρες που δεν θα πρέπει να αμφισβητηθούν για την ε, ιεράρχηση των αξιώσεων και επίσης θα πρέπει να επεκταθούν οι διατάξεις αυτές ώστε να ισχύουν και στις offline πωλήσει. Για να μην ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες μόνο για τις online πωλήσει. Όλα αυτά είναι ε, ανοιχτά ερωτήματα. Κύριε Αριμόν, πραγματικά δεν σας ζηλεύω καθόλου για, το, για τη δουλειά αυτή που έχετε μπροστά σας, γιατί θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Γιατί φαντάζομαι ότι τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη θεσπίσει ε, περαιτέρω κανόνες ε, δεν θα έχουν κανέν, καμία διάθεση να υπαναχωρήσουν. Και δεν καταλαβαίνω και γιατί θα έπρεπε να τους το ζητάμε αυτό. Ε, άρα ζητούμενο για μένα είναι ότι αν θέλουμε πλήρη εναρμόνιση θα πρέπει να γίνει αυτή με πάρα πολύ ε, υψηλές απαιτήσεις ή να υπάρξει μια ελάχιστη εναρμόνιση σε υψηλότατο επίπεδο ώστε να μην αρχίσουν τα κράτη-μέλη να νομοθετούν ε, διαφορετικά πράγματα από, από ό,τι ε, προβλέπει αυτή η πρόταση. Αλλά έτσι όπως έχει η πρόταση αυτή τη στιγμή η ομάδα μου, η πολιτική μου ομάδα δεν μπορεί να την αποδεχτεί. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, αν όχι να κάνω εγώ μερικά σχόλια. Κοιτάξτε, δεν θα αυξήσουμε το εμπόριο στην ψηφιακή ενιαία αγορά εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ισχυρή των καταναλωτών στο εμπόριο αυτό και οι καταναλωτές αν χάνουν σε υπάρχουσα προστασία καταναλωτών ε, ε, ή αν ε, τελούν συγχύσει ως προς τα δικαιώματά τους δεν θα έχουν εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά δικαιώματα εντός και εκτός διαδικτύου. Αυτό είναι κάτι το οποίο ψήφισε και το Κοινοβούλιο στην έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας ίσα δικαιώματα, υπάρχει το click and collect, υπάρχουν ε, και διάφορα είδη άλλων πολίσεων. Ε, το να χαθούν υπάρχοντα δικαιώματα και κτημένα όπως ε, το να τα έξι χρόνια να δίνουν δύο χρόνια για την επιστροφή. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά ε, αντίκειται πλήρως σε όλη τη δουλειά που κάνουμε στην κυκλική οικονομία. Ε, είναι σαν να λέμε ότι ε, ε, αυξάνεται το προσδόκιμο ε, ζωής και δεν λαμβάνεται αυτό υπόψη στην, στην, στην κοινωνία ε, με διάφορους τρόπους, ε, όταν δηλαδή δεν το βλέπουμε καθόλου μακροπρόθεσμα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην υπάρχουν πλέον τα ίδια δικαιώματα. Η αντιστροφή του, του άχθους απόδειξης είναι κάτι το καλό. Παρ' όλα αυτά κάποιες ενώσεις καταναλωτών ανησυχούν πάρα πολύ γιατί δεν υπάρχουν πολύ καλά δεδομένα που να προκύπτουν από την αξιολόγηση αντικτύπου. Το να πάμε στους μεγάλους ε, πολιτές ε, πλυντηρίων, smartphone, διαφόρων τέτοιων προϊόντων και να τους ρωτήσουμε πόσα πρώτα σας επιστρέφονται τους πρώτους δύο μήνες, έξι μήνες, τρία χρόνια, πέντε χρόνια. Είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Αν εγώ αγοράσω ένα καινούριο boiler στο σπίτι μου. Περιμένω να διαρκέσει πάνω από δύο χρόνια η ζωή του. Αν όχι θέλω να μπορώ να το επιστρέψω ή να το επιδιορθώσω. Αν δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια δουλειά που κινούμε τους, με τους πολιτές για να μπορούμε να καταλάβουμε τι είδους δεδομένα έχουν εκείνοι, τι στοιχεία έχουν εκείνοι, Υπάρχει περίπτωση να αυξήσουμε τελικά τις τιμές τους καταναλωτές με την αντιστροφή του άχθους απόδειξης. Δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο τον αντίκτυπο όλων όσων προτείνονται εδώ μπορεί να υπάρξει μία μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου και υπάρχει συνένεση μεταξύ της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων και ζητήσουμε περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία, αν αυτό πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε, τότε αυτό να κάνουμε. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και πάλι να απαντήσω εκείνα τα σημεία που έθεσαν πολλοί βουλευτές και αν έχω χρόνο θα απαντήσω και στα υπόλοιπα με μονομένα ερωτήματα. Το πρώτο που ρώτησαν πολύ, πέντε λεπτά αν είναι δυνατόν έτσι γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ε, θα προσπαθήσω τι να κάνω. Ε, το θέμα επιγραμμικών ή μη Σας είπα, συμφωνούμε απολύτως. Δεν θέλουμε να έχουμε διαφορετικούς κανόνες για το εμπόριο αυτό. Δεν θέλουμε ούτε να οδηγήσουμε σε σύγχυση τους πολίτες, τους καταναλωτές, ούτε να δυσκολεύσουμε τις επιχειρήσεις. Κάνουμε ε, την προσπάθεια REFIT ε, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θέλουμε τον Ιούλιο να έχουμε τα πρώτα στοιχεία, πολύ γρήγορα να ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση, να δημιουργήσουμε ομάδα ενδιαφερομένων. Το αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε. Αναλόγως των αποτελεσμάτων θα ληφθεί η απόφαση τι θα γίνει με τα αποτελέσματα αυτά. Πάντως η ιδέα θα μπορούσε να είναι είτε να μπει στην νομοθετική διαδικασία το αποτέλεσμα αυτό, είτε να κάνει μια νέα πρόταση τροποποιημένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε ακόμα και να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή προ όλε τι πολίτε. Το στρατηγικό αποτέλεσμα είναι δεν θέλουμε να είναι σε σύγχυση ο καταναλωτή, δεν θέλουμε να δυσκολεύουμε ε, περισσότερο τι επιχειρήσει και αυτό στο τέλο ε, μετράει και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Δεύτερο σημαντικότερο που ενδιαφέρει όλου είναι η προστασία των καταναλωτών και το επίπεδό τη. Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ σκληρά όταν κάναμε την πρόταση αυτή. Τι επιλογέ είχαμε. τι εξή τρει. βασικά. Είτε θα μέναμε στο επίπεδο του ελάχιστου κοινού παρονομαστή, που είναι περίπου το επίπεδο της οδηγίας πωλήσεων που έχουν όλες οι χώρες πάνω κάτω, είτε το άλλο ακρό θα ήταν να συλλέξουμε όλες τις ανώτατες μορφές προστασίας καταναλωτού από τα κράτη-μέλη. Εμείς επιλέξαμε την μέση εδώ, το αυξήσαμε σε ορισμένα σημεία, αλλά όχι παντού. Γιατί δεν το κάναμε, το είπαν πολλοί βουλευτές, γιατί δεν θέλουμε να μειώσουμε την εθνική προστασία των καταναλωτών, γιατί σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό επίπεδο, το ευρωπαϊκό αυξάνεται σημαντικά. Αλλά δεν θελήσαμε να μειώσουμε, γιατί φανταστείτε την κατάσταση αν λάβει όλες τι υψηλότερε προστασίε από όλα τα κράτη-μέλη, θα είμαστε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ε, σαφέστατα. Αλλά ποιος λιανέμπορο θα μπορούσε να πουλάει διασυνοριακά. Ε, τον ενθαρρύνουμε έτσι. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Ε, αναζητήσαμε τη μέση οδό λοιπόν που έχει το εξή πλεονέκτημα. Ε, υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για τις πωλήσει για να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή και ε, ανταγωνιστικές τιμές, έχοντας ταυτόχρονα πολύ ψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Για τα συγκεκριμένα, για τη διετία, για την εγγύηση, γιατί το επιλέξαμε αυτό. Διότι βασικά αυτό ε, έχει αποδειχθεί στην πράξη αποτελεσματικό. Ε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είδαμε και στοιχεία δεδομένα των καταναλωτών και είδαμε ότι μια σχετική πλειονότητα των καταναλωτών έλεγαν ότι η διετία για την εγγύηση είναι πιο λογική για τις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες προϊόντων που εξετάσαμε. Είπαν ότι είναι ένα λογικό ε, διάστημα για εγγύηση. Το δικαίωμα επιστροφής ή απόρριψης. Ε, το σκεφτήκαμε και αυτό. Τι κάναμε στην πρόταση. Στην ίδια την πρόταση θα έχουμε πιο εύκολη μετάβαση από το πρώτο επίπεδο στο δεύτερο επίπεδο ιεραρχίας για να τερματιστεί η σύμβαση σε σχέση με την οδηγία για τις πωλήσει. Και το δεύτερο υπάρχει και το δικαίωμα ε, ανάκλησης ή απόσυρσης που έχουμε 15 μέρες στην οδηγία ε, για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές κανονικά μέσα σε λίγες μέρες αποφασίσουν εφόσον έχουν βρει ένα ελάττωμα να αλλάξουν το προϊόν ή να το ε, επιστρέψουν. Ε, το πολύ πολύ μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει λοιπόν τεράστια διαφορά. Γι' αυτό κάναμε την πρόταση. Σε ό,τι αφορά το κρυφό ελάττωμα, βις κασέ, που προβλέπεται σε κάποιες χώρες ή ε, τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις του Ηνωμένο Βασίλειο, Αυτό το, το θέμα του κρυφού ελαττώματος τι σημαίνει. Χάνει την πρακτική του σημασία αν έχουμε διετία για την αντιστροφή του βάρους της απόφασης, ε, απόδειξη γνώμη. Διότι αυτό θα οδηγούσε μόνο για ελαττώματα που κανείς ανακαλύπτει μετά από δύο χρόνια. Και θα πρέπει ο πολιτής να ε, αποδείξει ότι υπήρχε ελάττωμα. Και δεν είναι πολλά τα προϊόντα. Πόσα είναι τα προϊόντα που μπορεί ε, να αποδείξουν οι καταναλωτές μετά από δύο χρόνια ότι το ελάττωμα ήταν από γεννησιμιού του προϊόντος. Άρα, αν έχουμε την αντιστροφή του βάρους απόδειξης, η διετία καλύπτει. Ε, τώρα, ε, τα ένδικα μέσα διατηρούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού, σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει αυτή η ρύθμιση, διότι η οδηγία δεν εναρμονίζει αυτό το στοιχείο. Και τώρα, να ε, έρθω στι συγκεκριμένε ερωτήσει πολλών ευρωβουλευτών. Κύριε Αριμόν γιατί όχι μία οδηγία αντί για δύο, βασικά για τους εξή δύο λόγου Πρώτον, αρχικά ήταν μία η οδηγία αλλά στο μεταξύ διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία αυτή ήταν πάρα πολύ μακροχρόνια και πάρα πολύ περίπλοκη και για λόγους νομοτεχνικούς το καλύτερο ήταν να σπάσει στα δύο. Ήταν πολύ περίπλοκη και κάθε φορά που είχαμε μια ιδιαιτερότητα του ψηφιακού περιεχομένου έπρεπε να ε, προβλέπουμε ειδικέ ρυθμίσεις που έκανε το όλο εγχείρημα πάρα πολύ ε, χρονοβόρο και δύσκολο να εφαρμοστεί. Και έχουμε και μια ρήτρα αναθεώρηση για το ψηφιακό περιεχόμενο, περιεχόμενο ακριβώς γιατί είναι ραγδαίε οι εξελίξεις, οι τεχνολογικές και εξελίξει στην αγορά. Ε, δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό για τις πωλήσει, μόνο για το ψηφιακό ε, περιεχόμενο, γιατί ούτε η αγορά αναπτύσσεται με τέτοιους ραγδαίους ρυθμούς και έχουμε και μεγάλη εμπειρία με την οδηγία για τις πωλήσει. Γι' αυτό τις πάσαμε στα δύο βασικά. Uh, Είπατε κύριε Άντερσον ότι η μελέτη αντικτύπου αφορά πολύ περιορισμένο μόνο αριθμό συνεντεύξεων. Έξι με μικρομεσαίες. Έχετε δίκιο. Απολύτως. Αλλά δεν είναι τα μόνα στοιχεία που έχουμε αυτά σε καμία περίπτωση. Κάναμε δύο ε, Έρευνε σε 20.000 περίπου επιχειρήσεις. Ευρύτατη δημόσια διαβόλευση πέρσι. Έχουμε ομάδα ενδιαφερομένων, ε, stakeholders που, που τη συμβουλευόμαστε ένα χρόνο ολόκληρο και εκτός αυτού είχαμε και κάποιες επιλεγμένες συνεντεύξεις σε μεγαλύτερο βάθος με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με εταιρείε που έχουν εμπειρία στο διασυνοριακό εμπόριο ακριβώς για να συζητήσουμε σε βάθος τις δικές τους εμπειρίες. Αλλά αυτό ήταν βασικά το κερασάκι στην τούρτα. Ε, είχαμε πολύ μεγαλύτερη, ευρύτερη διαβούλευση. Ε, αναφερθήκατε στο άρθρο 4, παράγραφος 3 για αποκλειστικά δικαιώματα. Αυτό ακριβώς είναι το ίδιο με την οδηγία για τις πωλήσει. Απλώς διευκρινίζει τα πράγματα, γιατί ως ο λιανικός πολιτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει στο καταναλωτή ότι μπορεί ένα προϊόν να είναι ελαττωματικό. Ε, αλλιώς δεν μπορείς να πουλήσει συγκεκριμένα είδη, αγαθά. Υπήρχε αυτό στην οδηγία των πωλήσεων, το καταλάβαμε και αυξάνει εδώ την προστασία των καταναλωτών, διότι τι λέμε, ότι αυτό γίνεται με δύο όρους και υποθέσεις, θα πρέπει να το γνωρίζει ο καταναλωτής και ρητά να το αποδέχεται. Αυτό δεν το έλεγαν τα προηγούμενα κείμενα η οδηγία των πωλήσεων, άρα το βελτιώνουμε αυτό το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Γιατί την κυρία Φανπόσοετ, ρωτήσατε για ε, την ε, ισορροπία αυτή και μπορεί να επιλέξει ο καταναλωτή επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Μα αυτό υπάρχει ήδη στην οδηγία για τι πωλήσει, αλλά στην πρόταση αυτή υπάρχουν όροι και προποθέσει που το περιορίζουν. Ε, όταν υπάρχει αδυναμία ή δυσαναλογία. Όταν είναι ένα αγαθό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί, γιατί είναι μοναδικό, δεν μπορεί να ζητήσει ο καταναλωτής να αντικατασταθεί ή όταν είναι δυσανάλογα δαπανηρό, κοινώ πανάκριβο, ε, μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση. Ε, παρακαλώ, ε, έχει περάσει η ώρα, κοινο πανακριβο μπορει να τελειώνετε. Ε, τότε σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Άλλες απαντήσεις μπορείτε να μας δώσετε γραπτός ή και online. Να ξαναπώ ότι για μας είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι κάνουμε κάτι που ε, βοηθά τους ε, καταναλωτές όταν έχουμε οργανώσεις των καταναλωτών που εκφράζουν ανησυχίες. Οπότε, με ενδιαφέρει πολύ τι θα κάνουν ο εισηγητής και οι σκιώδεις αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο όταν ε, λέμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και οι ίδιες οι καταναλωτικές οργανώσεις εκφράζουν ανησυχίε. Επόμενη συνεδρίαση 23 Μαΐου το απόγευμα στις 3 και μετά στις 24 ολόκληρη τη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη γραμματεία μας. Ah, Τους διερμηνείς και το προσωπικό που έμεινε μέχρι αυτήν την ώρα σήμερα το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.